Τώρα φτάνουμε ε, στην κοινή συζήτηση για το θέμα της περιφερειακής πολιτικής. Θα ήθελα λοιπόν να καλέσω ε, τις ε, εκθέσεις Λουχάν και Μανέσκου και θα δώσω το λόγο δίνοντας ε, καταρχήν στον κύριο Λούχαν ο οποίος έχει τέσσερα λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, Θέλουμε την έκθεση αυτή να απαντήσουμε στο ερώτημα του τίτλου. Αν είναι πραγματικά δυνατή η πραγματική εδαφική, κοινωνική και οικονομική ε, συνοχή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλλον αν είναι απαραίτητη για την ε, παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 271 οι περιοχές, περιφέρειες Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην πιο πλούσια από, αυτήν, αυτές ε, το ΑΕΠ είναι 334 φορές ψηλότερο από το μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ στην πιο φτωχή από αυτές ε, το ΑΕΠ της είναι 26% μικρότερο από το μέσο όρο. Ένα άλλο στοιχείο. Η οικονομική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ πιο αργή από αυτό την των ανταγωνιστών μας, των διεθνών μας ανταγωνιστών. Όπως ε, λέμε και στρατηγική Ευρώπη 2000, Ευρωπαϊκή Ένωση 2020, πρέπει να αναπτύξουμε στρατηγικούς τομείς και να δούμε και πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να γίνουμε πιο ισχυροί. Αντιμετωπίζουμε ένα δύσκολο έργο, γιατί ε, πέραν των αποτελεσμάτων της κρίσης ε, έχουμε και άλλες προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε. Για παράδειγμα, προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση, ε, δημογραφικές αλλαγές, κλιματική αλλαγή και όλα τα προβλήματα σχετικά με την ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια. Ο ρόλος της ε, πολιτικής συνοχής στην Στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση 2020 είναι αναμφισβήτητος. Η προτεραιότητα των πολιτικών μας θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τους στόχους της ε, στρατηγικής αυτής. Είναι απαραίτητη μια πολιτική συνοχή ανεξάρτητη με οι στόχοι της στρατηγικής μας θα επιτευχθούν μόνο αν αυξήσουμε τη συνέργεια ε, σε αποφενός και την συνοχή αφετέρου. Θα πρέπει να εφαρμόσουμε προγράμματα ε, πλατιά που θα καλύπτουν όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα δημιουργούν θέσει απασχόληση παντού και θα εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα όλων των περιφερειών. Θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στις ε, επενδύσεις στις υποδομές, υποδομές μεταφορών, τεχνολογίας πληροφοριών, επικοινωνίας, ε, έρευνας, ανάπτυξης, περιβάλλοντος, εκπαίδευσης Όλες αυτές οι υποδομές θα επιτρέψουν μεγαλύτερη προσβασιμότητα σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες και θα τους δίνουν ένα, μια ε, ίση, ε, κάποια ίσα δικαιώματα σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη του δυναμικού τους περιφερειακοί και τοπικοί στόχοι θα πρέπει να καθοριστούν με βάση τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής με δυνατότητα, ε, με, ανάλογα με τις ε, δυνατότητες παραγωγής προστιθέμενης αξίας κάθε μιας από αυτές. Θα πρέπει να γίνει αποκέντρωση στις τοπικές και περιφερειακές αρχές ε, για να διαχειριστούμε καλύτερα αυτή την πολιτική. Για να προάγουμε την οικονομική ανταγωνιστικότητα δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε το ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θα πρέπει να διαθέτουν ε, ενισχυμένη πρόσβαση στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση με καινούρια, και με καινούρια μέσα χρηματοδότησης. Η ενίσχυση ε, της, του αντικτύπου της πολιτικής συνοχής είναι απαραίτητη προκειμένου να υποστηρίξουμε την οικονομική ανταγωνιστικότητα. Εδώ θέλω να υπογραμμίσω την ανάγκη ε, απλοποίησης της χρήσης των κοινωτικών πόρων και ταμείων. Επίσης ε, θα πρέπει αυτά τα ταμεία να είναι πιο ευέλικτα, ε, θα πρέπει να διατηρήσουμε το ΑΕΠ ως βασικό κριτήριο για την επλεξιμότητα των περιοχών στο πλαίσιο της στρατηγικής συνοχής και τέλος είναι απαραίτητο η Κομισιόν να υποβάλει συγκεκριμένη πρόταση ό,τι αφορά την χρήση των ε, εταιρικών σχέσεων δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Για να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση πιο ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο, πιστεύω ότι ένα τμήμα των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής θα πρέπει να κατευθυνθεί προς την ε, υλοποίηση και τη διατήρηση την, ε, ενός ε, ρόλου ηγέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συγκεκριμένους ιδιαίτερα τομείς που η Ευρώπη έχει υψηλό δυναμικό. Η υλοποίηση της συνοχής εδαφικής, κοινωνικής και οικονομικής με επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς είναι απόλυτο απαραίτητη προπόθεση για να εξασφαλίσουμε την ανταγωνιστικότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε παγκόσμιο επίπεδο. Ευχαριστώ. Ε, ε, ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα τώρα να δώσω τον λόγο στον συγκεκριτή της δεύτερης έκθεσης την κυρία Μανέσκου. Έχετε τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως ξέρετε, η τωρινή παγκόσμια κρίση απαιτεί μια πάρα πολύ καλή διαχείριση και ειδικά στις, ε, στους τοπικούς φορείς οι οποίοι θα πρέπει να συνεταιριστούν για μια κοινή στρατηγική για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν ε, τα κονδύλια που είναι διαθέσιμα στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Η ιδιαίτερη σημασία της ε, κοινοτικής πολιτικής ε, για την ε, ευρωπαϊκή συνοχή θα πρέπει να γίνει συνείδηση όλων των κρατών μελών. Οπότε τοπική και περιφερειακή φορείς θα πρέπει να εμπλακούν ήδη από το προνομοθετικό επίπεδο για να έχουμε την καλύτερη εκμετάλλευση των μηχανισμών της ε, χρηστής ε, διοίκησης. Θα πρέπει λοιπόν ε, να παίξει αποφασιστικό ρόλο εδώ πέρα και η Κομισιόν. Η πρακτική αποδεικνύει είναι πιο αποτελεσματική η περιφερειακή πολιτική για την επίτευξη των στόχων αυτών. Άρα χρειαζόμαστε έναν κοινό ορισμό του όρου εταιρική σχέση. Και ζητήσαμε από την Κομισιό να επεξεργαστεί αυτόν τον ορισμό για να μπορέσουμε να έχουμε μια πραγματική τέτοια συνεργασία με τις ε, τοπικές αρχές. Αν λοιπόν βασιστούμε σε αυτές, αυτό θα έχει αποφασιστική σημασία για την πραγματοποίηση του ρόλου που μπορούν να παίξουν αυτοί οι φορείς ε, στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για περιοχές άστικες ε, της υπαίθρου και μεθοριακές. Επίσης, ε, δεν πρέπει να είναι αυτό αποτέλεσμα της ευρωπαϊκής κρίσης, αλλά να αποτελέσει γενικότερη αρχή της ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής. Δηλαδή, να χρησιμοποιήσουμε και να ενθαρρύνουμε το δυναμικό που υπάρχει σε αυτές τις περιοχές για το επόμενο για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού θα πρέπει να επεξεργαστούν προγράμματα με όλες αυτές τις ευρωπαϊκές περιφέρειες έτσι ώστε να δημιουργηθούν ή επιπλέον εκείνες προϋποθέσεις για να μην υπάρχει κανένα εμπόδιο στην χρηματοδότηση. Θα πρέπει λοιπόν να επεξεργαστούμε μια μικροπρόθεσμη πολιτική στόχευμένη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει τις ε, αρχές εκείνες, ε, τις τοπικές και τις περιφερειακές, να τις στηρίξει καλύτερα, αλλά βεβαίως και τις δραστηριότητες σε εθνικό επίπεδο. Στο πλαίσιο λοιπόν της ε, χρήσης αυτών των προγραμμάτων θα καταφέρουμε να παραμερίσουμε λάθη στον τομέα των δημοσίων προμηθειών. Θεωρούμε πως πρέπει να σταματήσει ο υπερβολικός έλεγχος. Έχουμε ζητήσει πάρα πολύ συχνά από την Κομισιόν να επεξεργαστεί οδηγίες για τις τυποποιημένους δημοσιονομικούς ελέγχους. Επίσης θα πρέπει εδώ πέρα να δούμε ποια θα είναι η συμμετοχή ιδιωτικών εταιριών όσον αφορά την ευρωπαϊκή συνεργασία. Να απευθυνθούμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τα μέλη της Επιτροπής συνεργαστήκαμε αρκετά καλά, έδειξαν αρκετά μεγάλη διάθεση για τη χρήση όλων αυτών των μέτρων για να αποτελέσει αυτό εγγύηση για το ότι τα μέτρα αυτά θα γίνουν δεκτά από την Κομισιόν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Uh, ευχαριστώ πολύ για την ακρίβειά σας και θα ήθελα να δώσω αμέσως το λόγο στον Ιωάννης Χάνα Καλώς ήλθατε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι βουλευτές, κυρία Μανέσκου, κύριε Λόχον, σας ευχαριστώ για τις δύο αυτές εκθέσεις σας, οι οποίες είναι επικοδομητικές και πάρα πολύ θετικές όσον αφορά την περιφερειακή πολιτική και νομίζω πως έρχονται και την κατάλληλη στιγμή δεδομένων το δεδομένη συζήτηση ε, που υπάρχει αυτή τη στιγμή για το μέλλον της ε, περιφερειακής ε, πολιτικής στο φόρουμ συνοχής που θα λάβει η χώρα τέλος Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου η πολιτική αυτή είναι μια πολιτική επενδύσεων στις περιφέρειες, στους ανθρώπους και βεβαίως θα πρέπει να είναι ορατή από τους ε, ανθρώπους και οπωσδήποτε Ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε προγραμματίσει 68 δισεκατομμύρια ευρώ για την καινοτομία στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο που θα βοηθήσουν ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να βοηθήσουν την ποιότητα της εργασίας, της μεθόδους παραγωγής, ε, την δυνατότητα προσφοράς υπηρεσιών. Και βεβαίως εδώ πέρα έχετε και οι δύο δίκαιο, πως ε, στο μέλλον η στρατηγική μας θα πρέπει να βελτιωθεί, να δούμε και τι θα γίνει με τους μελλοντικού ελέγχους ε, για να διασφαλίσουμε βεβαίως και τα οικονομικά συμφέροντα της κοινότητας αλλά να προσανατολιζόμαστε πολύ περισσότερο προς τα αποτελέσματα και βεβαίως κάτι το οποίο λέω πάντα και υπάρχει και στα συμπεράσματα να εστιαστούμε σε λίγες προτεραιότητες που αναφέρονται στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση 2020 ευελιξία στην εφαρμογή βεβαίως της διάφορης ε, περιφέρειες. Αυτά τα δύο δεν αποτελούν αντίφαση. Ειδικά το μέσο συνογή είναι πάρα πολύ σημαντικός για εμένα. Για εμένα είναι κάτι το ιδιαίτερα αγαπητό και νομίζω πως μπορούμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες ζωής στις περιφέρειες και να φροντίσουμε οι άνθρωποι να έχουν μια προοπτική στο μέρος στο οποίο γεννήθηκαν. Και αυτό είναι μια συνεισφορά στην ε, περαιτέρω ευρωπαϊκή συνεχή. Αυτό έχει μεγάλη σημασία και στην επόμενη προγραμματική περίοδο θα δούμε οπωσδήποτε το ρόλο των πόλεων. Ξέρετε πως 70% των Ευρωπαίων ζουν σε πόλεις, αλλά βεβαίως αυτό σημαίνει πως πρέπει να δούμε ιδιαίτερα τη σχέση πόλης πόλης-υπέθρου. Δεν πρέπει να μας ξεφεύγει αυτό Και εδώ πέρα βεβαίως θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αποφύγουμε τυχόν αλληλεπικάλυψη. Επίσης σημαντικό ήταν αυτό το οποίο ακούστηκε και συζητήθηκε εντό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δηλαδή όταν μιλάμε για τις περιοχές εκείνες με τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες και νομίζω πως αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το συναντάμε πάρα πολύ συχνά, δηλαδή το θέμα των δημογραφικών εξελίξεων στην Ευρώπη, όπου αφενός έχουμε αποψήλωση του πληθυσμού της υπαίθρου και από την άλλη μεριά έχουμε πάρα πολύ μεγάλη αστιφιλία. Οπότε πάρα πολλοί άνθρωποι συγκεντρώνονται σε ελάχιστο χώρο και από την άλλη, όπως σας είπα, έχουμε την ε, αποψήλωση της ε, υπαίθρου. Οπότε θα πρέπει να γίνουν επενδύσεις σε νέα και σε νέες και παλαιές υποδομές για να διασφαλίσουμε και την ανάπτυξη. Ιδιαίτερα σημαντικό αναφέρθηκε νομίζω ιδιαίτερα στην έκθεση της κυρίας Μανέσκου το θέμα της εταιρική σχέση, της συνεργασίας. Ναι, είναι σημαντικό να έχουμε μια πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, αλλά θα ήθελα ειδικά εδώ πέρα να σας πω πως είναι σημαντικό και οι περιφέρειες, το τοπικό επίπεδο να συμπεριληφθεί εδώ πέρα. Καμιά φορά έχω την αίσθηση όταν πηγαίνω στις περιφέρειες και το συζητάω πως ε, θα ήθελαν οι τοπικοί εκπρόσωποι να εκπροσωπούνται στο περιφερειακό επίπεδο και οι περιφερειακοί εκπρόσωποι στο εθνικό επίπεδο. Και δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Οπότε Βεβαίως πρέπει να σεβόμαστε το σύνταγμα της ε, κάθε χώρας, αλλά ε, σε μένα θα βρείτε έναν υποστηρικτή στο να μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε όλα τα επίπεδα και όλους τους ενδιαφερομένους, ε, ΜΚΟ και τα λοιπά, στα προγράμματα αυτά των επενδύσεων. Όσον αφορά τώρα τους οικονομικούς ελέγχους, θα επανέλθω νομίζω δεδομένου του ότι ήδη ξεπέρασα τον χρόνο μου. Θα επανέλθω στη δευτερολογία μου κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Σα Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστούμε και για το χαιρετισμό σας και τώρα θα περάσουμε στον γύρο των ομιλητών που μιλούν εξ ονόματος των διαφόρων κοινοβουλευτικών ομάδων. Καταρχάς για δύο λεπτά θα ακούσουμε τον κύριο Σιφ Μάτουλα από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα και εγώ να πω πως πρόκειται αυτή η περιφερειακή πολιτική είναι μία από τις σημαντικότερες και πιο επιτυχημένες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να υπάρχει μια συμμετοχή στην πολιτική συνοχής ε, και συμμετοχή στα διάφορα επίπεδα. Οπότε θα πρέπει να συγκεντρωθούμε σε αυτό και στο προσεχές ε, χρονικό πλαίσιο και να δούμε πώς θα επεξεργαστούμε την ε, πολιτική μας για να οδηγηθούμε στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020. Η έκθεση Μανέσκου τονίζει τον ρόλο τοπικών και περιφερειακών άρχων στο πλαίσιο της ε, πολιτικής ε, συνοχής. Επίσης, η έκθεση αυτή δείχνει πως αυτή η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση θα πρέπει να διευρυνθεί οριζόντια και αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουμε να εξαντλήσουμε το δυναμικό οικονομικής ανάπτυξης που έχουν οι περιφέρειες. Βεβαίω, όταν μιλάμε για περιφερειακή πολιτική θα πρέπει να έχουμε κατά νου τις ιδιότητες τοπικών και περιφερειακών διοικήσεων Οι διοικητικέ ικανότητε λοιπόν αυτές θα πρέπει να βελτιωθούν και να δημιουργηθούν χρηματοδοτικά μέσα τα οποία θα ε, επικαιροποιηθούν. Ο ρόλος λοιπόν δήμων και περιφερειών θα πρέπει να ε, ενδυναμωθεί, να έχουμε περιφερειακές εταιρικέ ε, σχέσεις δεδομένων των εξελίξεων της ανάπτυξης υπαίθρου για να αποκαταστήσουμε την ε, ισορροπία μεταξύ των διαφόρων ε, περιφερειών. Έτσι λοιπόν θα μπορέσουμε να έχουμε αυτό το αναπτυξιακό δυναμικό να το χρησιμοποιήσουμε και να τηρηθούν και οι τοπικές να τιμηθούν και να διατηρηθούν οι τοπικές ε, ιδιαιτερότητες. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια αποκέντρωση για να τα επιτρέψει όλα αυτά, η οποία δεν έχει επιτευχθεί πλήρως σε όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό σημαίνει πως πρέπει ε, ταυτόχρονα να έχουμε μια προσέγγιση η οποία θα σοχεύει στα αποτελέσματα. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω και να συγχαρώ και τους δύο εισηγητές για την συνεισφορά τους στην ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ συνάδελφε. Τώρα για δύο λεπτά έχει το λόγο εκ μέρου των σοσιαλιστών ο κύριος Κυρίλοφ. Ευχαριστώ. Θέλω να συγχαρώ ε, τις, τις, τους συναδέλφους για τις εξαιρετικές τους εκθέσεις. Ε, την κυρία Λούχαν και τον κύριο Μανέσκου. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι είναι σημαντικό ο ρόλο που έχει να διαδραματίσει η πολιτική συνοχή για την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών περιφερειών. Μιλώντα για τη συνέχιση τη πολιτική αυτή και των επιτευγμάτων τη, πρέπει να υπάρχουν οι επαρκεί πόροι. Σε καμία περίπτωση θα πρέπει να διατεθούν λιγότερα χρήματα για την πολιτική συνοχή σε σχέση με την παρούσα περίοδο προγραμματισμού. Κάτι άλλο που δεν επιθυμούμε είναι να υπάρξει επιπλέον ε, φόρτο για του δικαιούχου. Ο μελλοντικό σχεδιασμό τη πολιτική συνοχή βασίζεται στην απόφαση που θα λάβουμε από κοινού. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο με την πρόταση την οποία έχει διατυπώσει. Και γι' αυτό βασιζόμαστε και σε εσά, κύριε Επίτροπε Χάν, διότι ορισμένες από τις προτάσεις αυτές, όπως οι προποθέσει ε, ώστε να λάβουν τα κράτη-μέλη χρηματοοικονομική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά την άποψή μου χρειάζονται ε, κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες. Σε ό,τι αφορά τώρα τις περιφέρειες που χρειάζονται, πρέπει να ξέρουμε ότι οι περιφέρειες χρειάζονται υποστήριξη και δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε συνθήκες ε, ε, που θα τις οδηγήσουν σε προβλήματα λόγω τη ανεπάρκειας ορισμένων ε, κυβερνήσεων. Συμφωνώ λοιπόν κύριε Επίτροπο ότι είναι απαραίτητο αυτά τα επίπεδα να τα αναπτύξουμε. Είναι λοιπόν σημαντικό να μην αντικαταστήσουμε την αιρεσιμότητα και τις προϋποθέσεις, ε, να μην υποκαταστήσουμε λοιπόν με αυτή με την προϋπόθεση τα, τα άλλα προβλήματα που θέλουμε να διορθώσουμε. Ας επιτρέψουμε στις περιφέρειες να συμμετέχουν ενεργά. Ας τους επιτρέψουμε να νιώθουν ε, ότι έχουν την ιδιοκτησία αυτών των σχεδίων και προγραμμάτων. Ε, τις αφοδιάσουμε με τους απαραίτητους σπόρους και βέβαια να φροντίσουμε συγχρόνως να, να χρησιμοποιήσουμε τους σπόρους με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ Ευγένη, λέει ο Πρόεδρος, ε, εξ ονόματος των Φιλελευθέρων. Έχει το λόγο η κυρία Μάνερ και αυτή για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους δύο εισηγητές για τις δύο αυτές εκθέσεις οι οποίες νομίζω αποτελούν θεμέλιο για το μέλλον της ε, πολιτικής συνοχής και μια πολιτική συνοχή η οποία θα λειτουργεί είναι πάρα πολύ σημαντική για την ανταγωνιστικότητα. Πάντα βεβαίως λέγαμε πως η περιφερειακή πολιτική είναι πολιτική επενδύσεων και πράγματι αυτό πρέπει να γίνει και στο μέλλον. Με την ε, πολιτική αυτή συνοχής μπορούμε να ε, ανταποκριθούμε και στην ε, πρόκληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020 αν θέλουμε πράγματι να έχουμε βελτίωση της έρευνας και καινοτομίας και να αποτελέσει βεβαίως η πολιτική αυτή κομμάτι αυτών των στόχων. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τα πράγματα κάπως ευρύτερα. Γιατί η πολιτική συνοχή δεν είναι μόνο αλληλεγγύη Βεβαίως είναι λοιπόν θέμα και αλληλεγγύης αλλά και προώθησης της καινοτομίας. Κάτι το οποίο πρέπει να δούμε λοιπόν. Δηλαδή τουλάχιστον να έχουμε τα ίδια μέσα και στην επόμενη προγραμματική περίοδο όπως έχουμε αυτή τη στιγμή. Όπως ξέρετε η τέταρτη έκθεση η σχετική ανέφερε τους διάφορους παράγοντες για τους οποίους πρέπει να οδηγηθούμε προς μια κατεύθυνση που θα σχεδίσει τα αποτελέσματα. Κυρία Μανέσκο, εσείς αναφερθήκατε σε ένα θέμα κλειδί, δηλαδή το πώς μπορούμε να έχουμε μια καλή πολιτική σε όλα τα επίπεδα. Είχαμε κάποια αποτελέσματα τα οποία δεν ήταν τόσο ευχάριστα όσον αφορά παραδείγματο χάρη τα νούμερα της εφαρμογής. Θα πρέπει λοιπόν να το πάρουμε σοβαρά αυτό, να βρούμε μία λύση. Γι' αυτό θεωρώ πως η έκθεση Μανέσκου ε, είναι πάρα πολύ καλή ως προς αυτό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Μάνερ. Εκ μέρου των Πρασίνων έχει το λόγο για 1,5 λεπτό ο συνάδελφος Ζαν Πολ Μπεσέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. θα ήθελα να συγκεντρώσω την προσοχή μου στην έκθεση Λούχαν. Συμφωνούμε με τον κύριο Λούχαν, τουλάχιστον σε ένα σημείο, στο ότι οι πολιτικές αυτές, συνοχής, οι περιφερειακές, είναι κομβικές για την οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης, για μια κοινωνικά αρμονική ανάπτυξη, ισορροπημένη και αποτελεσματική περιβαλλοντικά έτσι ώστε τελικά να είμαστε ουσιαστικά ανταγωνιστικοί παγκόσμια. Ευχαριστώ τον εισηγητή γιατί δέχτηκε κάποιες από τις τροπολογίες μας οι οποίες δημιουργούν την αηφορία της οικονομίας, μιας οικονομίας με χαμηλή παραγωγή διοξιδίου του άνθρακα. Παρ' όλα αυτά δεν θα μπορέσουμε να υπερψηφίσουμε την πρότασή του γιατί το όραμα το οποίο αντιπροσωπεύει για την πολιτική συνοχή σαν αποκλειστικά μέσο παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας είναι κάτι το οποίο θεωρούμε ότι είναι περιορισμένο και ιδιαίτερα ανεπαρκές και στενό. Εμείς στην ουσία διαπιστώνουμε ότι ο εισηγητής στηρίζεται περίπου αποκλειστικά σε κάποια ποσοτικά στοιχεία τα οποία μεταφράζονται σε επίπεδο υποδομών ως κινητήριες δυνάμεις της ανάπτυξης. Όλο και περισσότερο. Αυτό είναι το βασικό του κριτήριο. Αυτό είναι κάτι το οποίο θεωρούμε ότι δεν είναι ε, αντίστοιχο των σημερινών αναγκών. Σημειώνει 246 λειτουργικά προγράμματα στην έρευνα και την ανάπτυξη και θεωρεί ότι αυτό είναι θετικό χωρίς να θέσει ερωτηματικά σχετικά με το περιεχόμενο των προγραμμάτων αυτών. Καλό είναι να ερευνά βέβαια κανείς, αλλά καλό είναι να ξέρει τι θέλει να ερευνήσει. Και δεύτερον, δεν θέτει ξεκάθαρους στόχους ο εισηγητής σε σχέση με... Πρέπει να ολοκληρώσετε κύριε Μπεσέτ. Λοιπόν, ο εισηγητής δεν ξεκαθαρίζει τα προγράμματά του. Εμείς θέλουμε πιο ξεκάθαρες επιλογές για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις τις οποίες αντιπροσωπεύει η επιλογή της πράσινης οικονομίας, του πράσινη New Deal, που θα είναι το μόνο που θα σπρώξει την Ευρώπη και τις περιφέρειές της προς τα πάνω. Ευχαριστώ κύριε Μπεσέ. Δεν βλέπω στην αίθουσα τον κύριο Ζόμπρο. Θα δώσω τώρα λοιπόν το λόγο στον κύριο Αγκουράκη, εξ ονόματος της Ενωτικής Ευρωπαϊκής Αριστεράς. 1,5 λεπτό κύριε Αγκουράκη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι εκθέσεις κινούνται στην ίδια αντιλαϊκή κατεύθυνση με τους στρατηγικούς σχεδιασμούς των μονοπωλιακών ομήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αστικών κυβερνήσεων που τους υπηρετούν. Διαχρονικά δεν υπήρξε κύριε Πρόεδρε και ούτε μπορεί να υπάρχει πολιτική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρά τις προσπάθειες να χρησιμοποιηθεί με στόχο την χειραγωγή των λαών. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαδεύεται από δύο βασικά στοιχεία το πρώτο είναι η βαθιά ανισομετρία που είναι σύμφυτο χαρακτηριστικό του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης και το δεύτερο βασικό στοιχείο της είναι ότι η διάθεση των κοινοτικών κονδυλίων δεν πάει για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών αλλά για έργα και υποδομές για την κερδοφορία του κεφαλαίου και ζεστό χρήμα για τους μονοπωλιακούς ομίλους μέσω από τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σήμερα σε συνθήκες εξέλιξης της καπιταλιστικής κρίσης ακόμα και αυτή η ψευδεπίγραφη αρχή της κοινοτικής αλληλεγγύης εγκαταλείπεται και αντικαθίσταται από την ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου. οι εκθέσεις και τα σχέδια των πολιτικών εκπροσώπων του κεφαλαίου για τη μελλοντική πολιτική συνοχής υπηρετούν τις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρηματικών ομήλων, την ταχύτατη προώθηση των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων της αντιλαϊκής στρατηγικής εε 2020 την άγρια επίθεση στα εργατικά ασφαλιστικά και κοινωνικά δικαιώματα της εργατικής τάξης. η ευρωπαϊκή ένωση και ο καπιταλιστικός τρόπος ανάπτυξης δεν είναι σε θέση να ικανοποιήσουν επίγουσες ανάγκες όπως η αντισυσμική προστασία η παιδεία και η υγεία και η πρόνοια. γι' αυτό το λόγο κύριε πρόεδρε η αποδέσμευση από την ευρωπαϊκή ένωση είναι περισσότερο ποτέ από ανάγκη σήμερα όπως και η πάλι για μια σχεδιασμένη σοσιαλιστική κεντρική ε, οικονομία. ευχαριστώ πάρα πολύ. Eh, Ευχαριστώ συνάδελφε. Κόλμαν ένα λεπτό. Πρόεδρε. Κανονικά θα έπρεπε να μιλήσει ο κ. Μπάφτον, ο οποίος όμως είναι αδιάθετος και θα ήθελα να παρουσιάσω τις απόψεις του. Όπως γνωρίζουμε, μαζί με την κοινή αγροτική πολιτική, τα περιφερειακά ταμεία είναι ένα μεγάλο τμήμα του κοινοτικού προϋπολογισμού. Για πάρα πολλά χρόνια ο Βρετανικό λαός είναι υποχρεωμένος να πληρώνει από την τσέπη του για προγράμματα που δεν τον ωφελούν καθόλου. Πρόσφατα, η υπηρεσία ερευνητικής δημοσιογραφίας έφερε στην επιφάνεια ότι αυτά τα προγράμματα χρησιμοποιούνται για να χρηματοδοτούνται βιομηχανίες πολεμικού τύπου, παραγωγής πολεμικών όπλων στην Ανατολική Ευρώπη. Υπάρχουν ενδυμικές εντωμεταξύ απάτες σε αυτό το κομμάτι του προϋπολογισμού και τα ταμεία δεν χρησιμοποιούνται και γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω από την κυβέρνηση συνασπισμού του Ηνωμένου Βασιλείου να, σταματήσει να πληρώνει πλέον και να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τους μη εγγεγραμμένους για 1,5 λεπτό κύριος Τσέγγεντη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η κατάσταση στην Ουγγαρία είναι ιδιαίτερη. Αν δείτε τις περιφέρειες που σχηματίζουν ένα συγκεκριμένο οικονομικό τμήμα και αν δείτε την ιστορία, αν δείτε το παρελθόν, θα δείτε ότι οι περιφέρειες αυτές ήταν μια ενότητα. Εμείς υποστηρίζουμε την παροχή βοήθειας αυτής στις περιφέρειες. Και θα πρέπει να καταργηθούν τα εμπόδια, οι φραγμοί που χωρίζουν τους Ούγγρους. Υπάρχει όμως κεντρική χρηματοδότηση και θα θέλαμε να απευθύνονται στις τοπικές κοινωνίες οι ε, πόροι αυτοί σε σχέδια για τα οποία είναι αρμόδιες τοπικές αρχές. Πρέπει λοιπόν ε, στόχος μας να είναι η περιφέρεια, το τοπικό επίπεδο, γιατί εκεί υπάρχει και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Είναι μια οικονομική ενότητα ουσιαστικά αυτές οι περιφέρειες. Είναι πιο λογικό λοιπόν να δίνουμε τους πόρους και ίσως και την εξουσία της αρμοδιότητας στο τοπικό επίπεδο. Επίσης οι κανονισμοί θα πρέπει να απλουστευθούν, οι ΜΜΕ θα πρέπει να συμμετέχουν στα σχέδια και οι περιφέρειες που υπολείπονται θα πρέπει να λάβουν βοήθεια για να ανακτήσουν το χαμένο έδαφος. Οι Βρυξέλλες όμως ε, αντί να δίνει εξουσίες ε, στις περιφέρειες ε, παίρνει, συγκεντρώνει εξουσίες όμως θα πρέπει στο προσκήνιο να μπουν πλέον οι περιφέρειες θα πρέπει να λαμβάνουν άμεση οικονομική ενίσχυση και έτσι θα ξεκινήσει και μια νέα εποχή και για όλες τις περιοχές Ουγγαρίας. Εδώ ολοκληρώθηκε ο γύρος των εκπροσώπων των πολιτικών ομάδων και τώρα θα περάσουμε στους υπόλοιπους ομιλητές με πρώτον για δύο λεπτά τον κύριο Όλμπριχτ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Λίγες είναι οι ευρωπαϊκές πολιτικές που προκαλούν τόσες ε, αντιπαραθέσεις ε, όσο η πολιτική συνοχής που θεωρείται από κάποιους ως ε, η κατεξοχήν σοσιαλιστική πολιτική, από άλλους όμως θεωρείται καπιταλιστική πολιτική. Κάποιοι θεωρούν ότι είναι δίκαιη η πολιτική, άλλοι πιστεύουν το αντίθετο. Υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν ότι η πολιτική αυτή ουσιαστικά καταργεί τις ε, διαφορές. Άλλοι πιστεύουν ότι ε, αυξάνει την ανταγωνιστικότητα. Η πολιτική αυτή όμως ε, ουσιαστικά είναι σχεδιασμένη για να αυξήσει τη συνοχή, για να προσφέρει μεγαλύτερη κοινωνική δικαιοσύνη στην Ευρώπη, για να προωθήσει τις καλύτερε και τι περισσότερε ευκαιρίε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα. Δεν υπάρχει λοιπόν αντίφαση και το λένε ξεκάθαρα αυτό και οι δύο εκθέσει. Στι εκθέσει αυτέ ε, τονίζονται κάποια στοιχεία που είναι σημαντικά και στη συζήτηση που διεξάγουμε εμεί σήμερα, αλλά και στη συζήτηση που αφορά το μέλλον τη πολιτική συνοχή. Στι δύο εκθέσει δίνεται έμφαση κυρίως στην εταιρική σχέση, στη σύμπραξη. Απευθύνομαι στον Επίτροπο. Σας παρακαλώ σκεφτείτε σκεφτείτε να συμπεριλάβετε ε, στη σύμβαση αυτή ανάπτυξης ένα αίτημα προς τα κράτη-μέλη, μια προϋπόθεση. Δηλαδή κάθε κράτος μέλος πριν την υπογραφή της Σύμβασης του Συμβουλίου να καθορίζει κατευθύνσεις, προτεραιότητες και βασικούς κανόνες. Και αυτό σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, τις περιφερειακές αρχές. Αυτό θα πρέπει να γίνεται σε εταιρική, στο πλαίσιο εταιρική σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορέσει πραγματικά να καταστήσει υπεύθυνα τα κράτη-μέλη για την εφαρμογή τη πολιτική συνοχή. Ευχαριστώ. Τώρα, ο κύριο Σταυρακάκη, έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Επίτροπε αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ και να ευχαριστήσω την εισηγήτρια κυρία Μανέσκου για την εξαιρετική συνεργασία και για το γεγονό ότι ήταν πάντα έτοιμη να συζητήσει και να λάβει υπόψη τι προτάσει συναδέλφων αναφορικά με το περιεχόμενο τη έκθεση. Σχετικά με το περιεχόμενο αυτή τη έκθεση που συζητάμε, είναι αδιαφυσβήτητο ότι η καλή διακυβέρνηση αποτελεί προπόθεση για την επιτυχία κάθε πολιτική, πόσο μάλλον για την πολιτική συνοχή που στηρίζεται στην αποκοινού διαχείριση και μεταβιβάζει το μεγαλύτερο μέρο τη ευθύνη για αυτή στι εθνικέ και περιφερειακέ αρχέ στις προκλήσεις που θέτει το περίπλοκο σύστημα αυτής της διαχείρισης η απάντηση είναι μία πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι αν λάβουμε υπόψη το μελλοντικό προσανατολισμό της πολιτικής συνοχής όπως τουλάχιστον διαφαίνεται έως κάποιο βαθμό στην πέμπτη έκθεση για τη συνοχή η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση τόσο στην οριζόντια όσο και στην κάθετη διάστασή τη θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην βιωσιμότητα των όποιων αναπτυξιακών πρωτοβουλειών και στην επιτυχία τη πολιτική. καλωσορίζω επίση το αίτημα για περαιτέρω απλούστευση των κανόνων καθώ και για μεγαλύτερη τεχνική υποστήριξη των τοπικών αρχών από πλευρά τη ευρωπαϊκή επιτροπή ω παράγοντε που θα διασφαλίσουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή δυνητικών δικαιούχων στα προγράμματα και στην απορρόφηση πόρων κατά βιώσιμο τρόπο μέσα από τι αξιολογήσει που διεξάγει πλέον η ευρωπαϊκή επιτροπή. έχουμε στοιχεία για το ποιοι φορεί παρουσιάζουν σταθερά προβλήματα σε σχέση με τη διοικητική του ικανότητα στην υλοποίηση προγραμμάτων πολιτική συνοχή. όπω επισημαίνεται και στην έκθεση η πρόσθετη τεχνική βοήθεια προ αυτού του φορεί σε συνδυασμό με την ενίσχυση τη πρωτοβουλία train the trainers τη ευρωπαϊκή επιτροπή θα διασφαλίσουν την ενίσχυση τη διοικητική ικανότητα ακόμα και των πιο μικρών φορέων σε τοπικό επίπεδο τέλος η μεγαλύτερη ενοποίηση και εναρμόνιση των κανόνων των διαθροτικών ταμείων πιστεύω ότι θα συμβάλει καθοριστικά στις προσπάθειες απλοποίησης και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφε. Για δύο λεπτά η κυρία Χιουσμενόβα. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ συνάδελφε. Εδώ και λίγες μέρες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε το πρόγραμμα δράσης για τη στρατηγική του 2020. Και γι' αυτό θα ήθελα να εξετάσω την έκθεση Λούχαν μέσα από αυτήν την ψηφοφορία, μέσα από αυτήν την απόφαση. Θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι στην έκθεση αυτή διαμορφώνεται ένα πλαίσιο για την πολιτική συνοχής. Αυτή η πολιτική παίζει σημαντικό ρόλο στην ανταγωνιστικότητα της Ένωσης. Σίγουρα με την στρατηγική αυτή η παραδουνάβιο στρατηγική αποτελεί ήδη ένα τέτοιο πλαίσιο αντίστοιχο με την βαλτική στρατηγική. Όλα τα μέτρα λοιπόν τα οποία θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας έχουν πολύ μεγάλο ρόλο να παίξουν. Σαν παράδειγμα ζητείτε να υπάρξει μεγαλύτερη δυνατότητα σύνδεσης με άλλες περιοχές και εδάφη στα πλαίσια αυτής της πολιτικής συνοχής. Αυτό έχει μεγάλη σημασία και είναι κάτι που θα πρέπει να χαρακτηρίσει όλες τις επιμέρους στρατηγικές πολιτικές ανάπτυξης όπως την Παραδουνάβιο. Και επίσης θα πρέπει να υπάρξει ειδική προσπάθεια για τις περιοχές στις οποίες σημειώνεται μια σημαντική καθυστέρηση. Η έκθεση νομίζω κάνει επίσης και μια σωστή σύγκριση ανάμεσα στις διαφορετικές πλευρές που αποτελούν την πολιτική αυτή και οι οποίες θα παίξουν σημαντικότερο ρόλο από ό,τι σήμερα στο μέλλον. Σας ευχαριστούμε κυρία Χιουσμένοβα. Τώρα για δυόμιση λεπτά έχει το λόγο η κυρία Σρέντερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους εισηγητές για την ορθή διακυβέρνηση, ειδικά για την καλή συνεργασία και τους συγχαίρω για αυτή την καλή έκθεση έκθεση η οποία νομίζω δείχνει στην Κομισιόν τι πρέπει να γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα, ειδικά όσον αφορά την αρχή της ε, ε, εταιρικής σχέσης. Λέει πως θα πρέπει να συμπεριληφθεί το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και οι κοινωνικοί φορείς και οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών σε όλες τις φάσεις των διαρθρωτικών ταμείων και στην αξιολόγηση αυτό σημαίνει υποχρέωση δηλαδή των κρατών μελών να οδηγηθούν σε μια πραγματική εταιρική σχέση, να δώσουν εξουσίες σε αυτούς τους εταίρους, να μπορούν να μιλάνε ως ίση προς την διοίκηση και να έχουν πραγματική επιρροή στη διαμόρφωση των προγραμμάτων. Δυστυχώς μέχρι τη η Κομισιόν δεν δείχνει καμία τέτοια όρεξη. Αυτό ε, ισχύει και για την τρέχουσα περίοδο και φαίνεται από τις προτάσεις που έκαναν και χαιρετίζω αυτό το οποίο υπόθηκε πως εάν ε, καταλήξουμε σε αυτή την σύμβαση. Κάτι τέτοιο θα είναι δυνατόν μόνο εάν υπάρχει εταιρική σχέση και οι εταίροι θα μπορούν να συμμετέχουν επί ίσης όρης στην ανάπτυξη αυτών των σχεδίων. Αλλιώς υπάρχει ο κίνδυνος από μια Ευρώπη των περιφερειών να πάμε σε μια Ευρώπη των κρατών μελών και δεν μπορεί να είναι αυτός ο στόχος μας. Στόχος μας είναι η περιφερειακή ανάπτυξη και η συμμετοχή του τοπικού και περιφερειακού επίπεδου των εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών. Ευχαριστώ. 1,5 λεπτό επίσης για τον κύριο Φερέιρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ανισότητες σε περιφερειακό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο και εντός των χωρών και μεταξύ των χωρών και αυτό συνιστά σαφή αποτυχία του στόχου της συνοχής. Η πολιτική συνοχής δεν είναι μια πολιτική η οποία είναι απομονωμένη από τις λοιπές πολιτικές. Υπηρεάζεται αλλά και επηρεάζει τους πολιτικούς προσανατολισμούς αλλά και γενικότερα σε μακροοικονομικό επίπεδο. Επηρεάζει τους μισθούς. Βλέπουμε ότι οι δημόσιες υπηρεσίες ε, υποβαθμίζονται Γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει κάποιε οικονομικέ πολιτικέ, ε, όμω οδηγεί τελικά στην αύξηση τη στόχα και τη ανεργία, απομακρύνοντα όλο και περισσότερο από το στόχο τη συνοχή. Η πολιτική συνοχή φυσικά και δεν ε, αντιστάθμισε τι ανισορροπίε από την ένταξη στην ε, ενιαία αγορά από την ΟΝΕ διότι έχει οδηγήσει σε τελείως διαφορετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Επίσης δεν είναι επαρκής η πόρη της συνοχής και η οικονομικοί πόροι ουσιαστικά δεν βασίζονται στην πραγματική αλλά σε μια ονομαστική σύγκληση και αυτοί είναι οι λόγοι, αυτά είναι τα σφάλματα τα οποία θα πρέπει να διορθωθούν. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τη συνοχή, θα πρέπει να αλλάξουμε τι μακροοικονομικέ πολιτικέ, θα πρέπει να στηρίξουμε την παραγωγή, την ανάπτυξη των παραγωγικών ικανοτήτων κάθε χώρα, κάθε περιφέρεια. Θα πρέπει να προωθήσουμε το δυναμικό της κάθε χώρας, τους ίδιους πόρους. Θέλουμε ε, απασχόληση, ενίσχυση της κοινωνικής υποστήριξης των δημόσιων υπηρεσιών για να έχουμε ε, την αποτελεσματική οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή. Τώρα ο συνάδελφος Σκοτά έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η έκθεση Μανέσκου. Νομίζω ότι οι πολιτικές συνοχές θα κερδίσουν πολλά από μια σωστότερη διακυβέρνηση και μια καλύτερη ε, θα έλεγα κατανομή των ευθυνών σε όλα τα επίπεδα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί κάποιες πρωτοβουλίες οι οποίες θα πρέπει να αναλυθούν και σε επίπεδο τοπικό και περιφερειακό. Και σε αυτό το επίπεδο πρέπει να υπάρξει σωστό συντονισμό των κοινοτικών προγραμμάτων. Η συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο θα πρέπει να είναι διαφανής και να επιτρέπει την ισότιμη συμμετοχή όλων των οντοτήτων που συμμετέχουν. Και πρέπει να υπάρξει και σωστή ενημέρωση σε επίπεδο υποεθνικό σε εισαγωγικά μέσα από πρωτοβουλίες όπως το Εράσμους και γι' αυτό θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ θα επιτρέψει να υπάρξουν και ανταλλαγές χρηστών πρακτικών για να βελτιώσουμε την διαχείριση των περιφερειακών ταμείων. Δύο λεπτά τσέλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε αγαπητοί συνάδελφοι. Πρώτα απ' όλα λυπούμε για το ότι πάλι μια φορά μια σημαντική έκθεση για τη συνοχή βρέθηκε στο τέλος της ημέρας. Δεν ε, ανταποκρίνεται αυτό στην ε, πολιτική σημασία της πολιτικής συνοχής. Ευχαριστώ λοιπόν τους δύο συγητές οι οποίοι μας δείχνουν ε, σε ποιο βαθμό ήταν επιτυχημένη η Ευρωπαϊκή Ένωση στην πολιτική συνοχής και για το τι πρέπει να συνεχίσει. Και βεβαίω αυτό σε ένα πολιτικό σύστημα πολυεπίπεδο. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν γίνεται άμεσα αντιληπτή από τους πολίτες η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έργα υποδομής, με στήριξη της κοινοτομία, ε, της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης της περιφέρειας. Στην τωρινή συζήτηση για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέρα από τα νομίσματα και τα οικονομικά, πρέπει με την ίδια έντοση να γίνει η συζήτηση για το τι χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση για την εσωτερική της συνοχή για να μην υπάρχει έτσι αυτή η απομάκρυνση των περιφερειών και άλλα μετά των κρατών μελών. Βλέπουμε πως υπάρχει νέος ανταγωνισμός στην παγκόσμια αγορά και άρα χρειαζόμαστε περισσότερες κοινέ δυνάμεις και περισσότερη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε αυτό σημαίνει πως θα πρέπει η πολιτική συνοχής να προσανατολιστεί στα έργα εκείνα τα οποία ωφελούν συνολικά την Ευρώπη που δίνει τη δυνατότητα στα κράτη να παραμείνουν ισχυρά και στα στενέστερα κράτη να γίνουν ισχυρά. Μου φαίνεται λοιπόν πέραν από τους τωρινούς στόχους να υπάρχει μεγαλύτερη αίρεσιμότητα και να στραφούμε περισσότερο παραδείγματο χάρη στην καινοτομία και στην έρευνα, στην συγκοινωνία και στην ε, ενέργεια. Επίσης, νομίζω πως είναι απαραίτητο αυτό το οποίο λέει η Κομισιόν, δηλαδή να δημιουργηθεί ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο για να υπάρχουν εκείνοι οι εταίροι ανάπτυξης μεταξύ κρατών μελών, κομισιών και τοπικών εκπροσώπων. Αυτό σημαίνει όμως πως οι τοπικές αρχές θα πρέπει να μπλέκονται στη διαδικασία αυτή όσο το δυνατόν νωρίτερα. Κύριε Τσέλερ, παρακαλώ ολοκληρώστε. Για να έχουμε λοιπόν πραγματική πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέξτε μου ακόμη μια παρατήρηση για τον κύριο Κόλμαν, ο οποίος δυστυχώς έβγαινε πνεύσα. Να υπενθυμίσω, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ελεύθερη ε, ναι, ένας ελεύθερος συνεταιρισμό κρατών. Όποιος θέλει να φύγει μπορεί να φύγει. Αλλά δεν ξέρω εάν οι πολίτες ε, Σκοτίας, ε, Ουαλίας, Βόρειας Ιρλανδία και Αγγλίας θέλουν να κάνουν κάτι τέτοιο. Σα ευχαριστώ. Δεν βλέπω τον κύριο Γκάλεχερ στην αίθουσα. Επομένω, θα δώσω το λόγο στην αγαπητή κυρία Ματσόνη, η οποία έχει δύο λεπτά για την παρέμβασή τη. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπο, βάζουμε τις βάσεις για την Ευρώπη του 2020, μια Ευρώπη καινοτόμο, μια Ευρώπη έξυπνη, μια Ευρώπη όμορφη. Για να τα πετύχουμε όλα αυτά πρέπει να δώσουμε τον αγώνα της ανταγωνιστικότητας και να τον κερδίσουμε. Η πολιτική συνοχή στα πλαίσια των τριών πλευρών της, δηλαδή την εδαφική, την κοινωνική Κοιτάξτε, παρακαλώ να σκεφτείτε ότι λέει ο πρόεδρος ότι σας διαμηνεύουν ε, ε, από τις υπηρεσίες διαμηνίας και παρακαλώ να επιβραδύνετε. Λοιπόν, πιστεύω ότι είναι το μέσο στο οποίο θα πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας. Δεν νομίζω ότι εδώ στον τομέα αυτό μπορούμε να προχωρήσουμε σε περικοπές. Νομίζω ότι θα πρέπει να εφαρμόσουμε σωστότερα την πολιτική συνοχή σε εκεί όπου δείχνει να έχει αδυναμίες. Επί τη βάση της ανάλυσης των αποτελεσμάτων, η Αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή με την έκθεση Λιούχαν δείχνει τη σχέση που έχει η ανάπτυξη με την συνοχή και δείχνει και ποιες πιθανώς μπορεί να είναι οι διορθωτικές ενέργειες εφόσον η Ευρώπη μπορέσει να ξεπεράσει τις περιφερειακές ανισότητες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο που δέχτηκε την τροπολογία που είχε καταθέσει σχετικά με τις ευνοϊκές ε, φορολογικές ρυθμίσεις για μεταβατικές περιόδους μέχρι πέντε ε, χρόνια όπως είχαμε αποφασίσει και παλαιότερα το 2006. Νομίζω ότι είναι ένας τρόπος για να διορθωθούν τα προβλήματα της πολιτικής συνοχής όπως η γραφειοκρατία, η ανεπάρκεια ταυτόχρονα ελέγχου και για όλα αυτά τα μεθοδολογικά προβλήματα προτείνεται να υπάρξουν διορθωτικές ενέργειες για την βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων αυτής της πολιτικής. Όπως υπογραμμίζει η έκθεση Λούχαν, θα πρέπει εμείς να ζητήσουμε τη βελτίωση της εταιρικής σχέσης σε οριζόντιο κάθετο επίπεδο των τοπικών αρχών της κεντρικής διοίκησης του ιδιωτικού τομέα και να βοηθήσουμε επίσης την πρόσβαση στην χρηματοδότηση και την απλούστευση των διαδικασιών και ταυτόχρονα να παρατείνουμε την διατήρηση των μεταβατικών διατάξεων ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο κρίσης. Αυτό θα βοηθήσει την ανάπτυξη ξεβόμενη πάντα τις περιφερειακές ειδικέ συνθήκες. Υπογραμμίζω σε δύο τομείς την καινοτομία και τις υποδομές. Λοιπόν, έχει σημασία η έκθεση αυτή γιατί μας επιτρέπει όλους μας να έχουμε μπροστά μας ένα σωστό τρόπο για να μπορέσουμε να πετύχουμε τον στόχο τον οποίο έχει τον τίτλο η έκθεση. Σα ευχαριστώ. Θέλω να σα πω το εξής. Επειδή είμαι υπεύθυνο στο Προεδρείο για τα θέματα μετάφραση και διερμηνία, θα ζητήσω από τι υπηρεσίε του ημικυκλίου να μου αναβοσβήνει ένα φω κάθε φορά ε, που να το βλέπετε κι εσείς γιατί μου το λένε ότι δεν πρέπει να συνεχίσει ο μιλητής αλλά ίσως καλό θα ήταν και σε εσά, στο έδρανο το καθένα σα μπροστά του να έχει ένα φω που να αναβοσβήνει, που να του λέει ότι πάει πολύ γρήγορα και δεν ε, μπορούν να τον ε, μεταφράσουν οι διερμηνεί. Θα μεταφέρω λοιπόν την ε, αναγκαιότητα αυτή. Δεν έχει καμία σημασία να αναβοσβήνει το κουμπί στο Προέδρου το έδρανο που είναι ο διαμεσολαβητής ουσιαστικά. Καλό θα ήταν και ο μιλητή να το βλέπει όταν μιλάει πολύ γρήγορα. Λοιπόν, τώρα για δύο λεπτά έχει τώρα το λόγο ο κύριο Τεσέιρα. E- Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θέλω να συγχαρώ τους συναδέλφους Λούχαν και Μανέσκου για τις εκθέσεις τους. Συμβάλλουν τα μάλα στη συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή για τη νέα πολιτική συνοχής για τα έτη από 2014-2020. Η πολιτική, ε, οικονομική, κοινωνική και δαφική συνοχή είναι πολύ σημαντική για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό θα το πετύχουμε αν συνειδητοποιήσουμε ότι μόνο αν ενισχύσουμε την περιφερειακή διάσταση θα μπορούμε να έχουμε συνοχή στο εσωτερικό της ε, Ευρώπης και ανταγωνιστικότητα για προς το εξωτερικό. Να τονίσω κάποιες πτυχές. Πρώτα απ' όλα, αποκέντρωση. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές ε, και κυρίως οι τοπικές αρχές που συμμετέχουν περισσότερο και συμβάλλουν περισσότερο στην εφαρμογή της πολιτικής συνοχής θα πρέπει τα κράτη-μέλη να ζητούν από τις τοπικές αρχές να συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις επίσης όρες με τους εθνικούς εκπροσώπους. Και Επίσης, ενίσχυση του ρόλου των τοπικών και περιφερειακών αρχών για την εποπτεία και την διαχείριση των προγραμμάτων. Μόνο με αυτόν τον τρόπο, μόνο με τη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης σε όλα τα επίπεδα θα γίνει σεβαστή και η αρχή της επικουρικότητα. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι να έχουμε μια πιο απλή αρχιτεκτονική. όχι λόγω της οικονομικής κρίσης, αλλά πρέπει να ισχύει και στο μέλλον για να υπάρχει χρηστή εφαρμογή της πολιτικής συνοχής. Στόχος της Λισαβόνας ήταν η προσέγγιση των πολιτών. Δεν θα πρέπει να στην Ευρώπη. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε όχι μόνο αυτό, αλλά να αποφύγουμε να είναι πολύπλοκα τα συστήματα, να είναι αποτρεπτικά για να μην συμμετέχουν οι πολίτε. Πρέπει να είναι πιο απλά τα πράγματα. Έτσι θα καταφέρουμε τη μεγαλύτερη εδαφική συνοχή και έτσι θα εξαλείψουμε τι ανισότητε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι θα μειώσουμε το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών περιφερειών. Πρέπει βέβαια να υπάρχει, όπως καταλαβαίνετε, και μεγαλύτερη ευθύνη. Αυτή την ευθύνη όλοι την μοιραζόμαστε. Έτσι θα έχουμε μια πιο ισχυρή και πιο ανταγωνιστική Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βίγκλερ για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τους δύο εισηγητές και να ευχαριστήσω ειδικά τον Πετρολούχαν για αυτό το οποίο είπε για τη μελλοντική στρατηγική από το 2014 και μετά. Αν και βεβαίως ε, τα συμπεράσματα για την ε, πέμπτη έκθεση είναι ακόμα πρώτες ιδέες στην Κομισιόν, νομίζω πως η έκθεση του συναδέλφου είναι μια καλή αρχή της τοποθέτησης του Κοινοβουλίου έναντι της ε, Κομισιόν. Επίσης θεωρώ σωστό η πολιτική συνοχής ε, να συνδεθεί με την στρατηγική 2020 θα πρέπει όμως να συνεχίσουν οι περιφέρειες να μπορούν να θέτουν προτεραιότητες. Δεν είναι ίδιες όλες οι περιφέρειες και ούτε όλα τα κράτη-μέλη. Δύο, τρεις το πολύ προτεραιότητες ε, θα πρέπει να εφαρμοστούν λέτε. Αυτό δεν σημαίνει όμως εδώ πέρα πως έχουν τον απαραίτητο χώρο που χρειάζεται για να κινηθούν οι περιφέρειες. Θα πρέπει να μπορούν να διαλέξουν. Παραδείγματο χάρη να δούμε τις ιδιαιτερότητες όπως οι δημογραφικές εξελίξεις οι οποίες μπορεί να μην ληφθούν υπόψη ε, ειδικά όσον αφορά τις ανάγκες των ε, περιφερειών οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για τα οποία δεν λέει πάρα πολλά η Κομισιόν. Επίσης θα πρέπει να πω πώ δεν επιτρέπεται να εξασθενήσουν οι περιφέρειες έναντι των ε, κρατών μελών. Βλέπετε πως οι περιφέρειες έχουν τελείω διαφορετική διάσταση και ρόλο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να του αποδείτε η ανάλογη σημασία. Οπότε θα πρέπει να δουν ποιε θα είναι οι εξελίξει και οι καινοτομίε στις εταιρικέ σχέσεις μεταξύ Κομισιών και κρατομελών. Να αφαιρθώ επίσης στον ε, στόχο 3 συμφωνώ με τον συγητή όταν μιλάει για τις μεθοριακές περιοχές, ειδικά στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ πέρα πρέπει να το δούμε αυτό. Νομίζω πως ε, δεν δίνεται αρκετή σημασία στις περιοχές αυτές ε, όσον αφορά τη μελλοντική ε, διαμόρφωση αυτής της πολιτικής. Ειδικά δεν στην πατρίδα μου τη Σαξονία πολλά μπορεί να γίνουν ακόμα. Δύο λεπτά κυρία Ματέρα. Τα στοιχεία που δίνει το ελεγκτικό συνέδριο στα πλαίσια της ετήσιας έκθεσης ε, από το 6 μέχρι το 2008 για τα συστήματα ελέγχου διαχείρισης των περιφερειακών ταμείων είναι ανησυχητικά. Τα συστήματα ελέγχου δεν ήταν καθόλου ικανοποιητικά και έφταναν σε ένα επίπεδο αναγνωρισμένου λάθους 12% το 2006 και 11% το 2008. Πρέπει να μειώσουμε αυτό το ποσοστό λάθος. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσει τον ελεγκτικό της ρόλο σε επίπεδο τοπικό και περιφερειακό η επεξεργασία ενός σωστού οδηγού για τη συμπεριφορά των ιδιωτικών αλλά και δημοσίων ή δημοτικών εταίρων και στοιχεία, συμβουλές για το πώς θα πρέπει σε πολυεπίπεδο ε, τρόπο να εφαρμοστούν όλες αυτές οι συστάσεις θα βελτιώσουν την περιφερειακή μας πολιτική. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να βοηθήσουν τις τοπικές αρχές, ιδιαίτερα μετά από τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Θα πρέπει να διευκολύνουμε τη συνεργασία σε επίπεδο διαμεθοριακό, γιατί σε πολλές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δυναμικό το οποίο μπορεί να εκμεταλλευτεί κανείς σε επίπεδο συνεργασίας ανάμεσα σε περιφέρειες γειτονικών κρατών μελών είναι υψηλότατο. Ιδιαίτερα σε τομείς όπως ο τουρισμός, η γεωργία, η βιομηχανία και οι περιβαλλοντικές πολιτικές. Εδώ θα ήθελα να πω, μια και δεν καθυστεύσω, να χαιρετήσω του διερμηνείς οι οποίοι κάνουν εξαιρετική δουλειά. Σας ευχαριστώ και κυρίω γιατί μιλήσατε σε ένα πολύ ωραίο ρυθμό. Και έτσι δεν είχαμε προβλήματα με τους ε, διερμηνείς που πράγματι ενίοτε δεν μπορούν να παρακολουθήσουν την ταχύτητα. Τώρα για δύο λεπτά θα ακούσουμε τον κύριο Κοσλόφσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Καταρχάς θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η έκθεση αυτή θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική και θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή, τον κύριο Λούχαν, για την εξαιρετική δουλειά που έκανε. Νομίζω ότι η πολιτική συνοχή πρέπει να είναι μία από τις βασικές πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολιτική εχμής. Θα πρέπει ως οριζόντια πολιτική να καθορίζει τις κατευθύνσεις των τομεακών πολιτικών και να οδηγεί σε βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών περιφερειών και να ενισχύει την παρουσία της Ευρώπης στις παγκόσμιες αγορές. Θα πρέπει να υπάρξει ένα ευέλικτο μοντέλο για την πολιτική συνοχή. Με αυτό το ε, πολυεπίπεδο μοντέλο θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε να πάνε και σε άλλες περιφερειές ε, και τοπικές και σε άλλα τοπικά επίπεδα οι πόροι των ε, διαθετικών ταμείων. Ήμουν υπεύθυνο σε μια περιφέρεια 20.000 κατοίκων ε, για τα, μέσα, για τα μέσα συνοχής, των μηχανισμούς συνοχής, βάσει του συγκεντρωτικού και του αποκεντρωμένου μοντέλου, δηλαδή επιχειρησιακά περιφερειακά προγράμματα για την περίοδο 2007-2013. Έχοντα εμπειρία λοιπόν, μπορώ να πω με κάθε βεβαιότητα ότι το αποκεντρωμένο μοντέλο είναι πολύ καλύτερα προσαρμοσμένο για να αξιοποιήσουμε το δυναμικό στο τοπικό επίπεδο και να έχουμε θετικές, ε, θετικά αποτελέσματα. Είμαι πεπισμένος ότι θα πρέπει αποφάσεις να λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά ο τρόπος επίτευξης των στόχων με βάση τις αποφάσεις και σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας θα πρέπει να γίνεται στο πλέον ε, στο καλύτερα προσαρμοσμένο επίπεδο, δηλαδή στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, στο περιφερειακό και στο τοπικό επίπεδο. Είναι επίσης απαραίτητο να συνδεθούν οι δαπάνες με τους επιδιωκόμενους στόχους. Η δημιουργία θέσεων εργασίας και κοινωνική ένταξη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Εδώ ολοκληρώθηκε ο γύρος των γεγραμμένων ομιλητών και θα περάσουμε στη διαδικασία της προσέλκυσης της προσοχής του Προέδρου. Catch the Eye. Μετά το ένα λεπτό να ξέρετε ότι θα κόβω αυτομάτως το μικρόφωνο. Η κυρία Ελένα Μπατσέσκου είναι η πρώτη ομιλήτρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Λούχαν για την έκθεση αυτή. Είναι ε, έκθεση με μεγάλη σημασία και για την ε, Ρουμανία. Κατά την άποψή μου η στρατηγική 2020 θα πρέπει να αποτελέσει ένα σχέδιο αηφόρου ανάπτυξης ε, για να έχουμε μη... Γι' αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να υπάρχει μια καλύτερη παρουσία προς τα έξω για να έχουμε και βεβαίως αποτελεσματικότερη εργασία στο εσωτερικό επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημαντικό ρόλο παίζει εδώ πέρα η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των περιφερειών σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα μέσα χρηματοδότησης ε, για τα επενδυτικά αυτά έργα είναι πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Η Ρουμανία τώρα και στο διάστημα μετά το 2014 αναμένει πάρα πολλά κονδύλια. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μπασέσκο. Κύριος Άλβης έχει τώρα το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αναγνωρίζουμε τη σημασία που έχει η πολιτική συνοχής στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ανάπτυξη της σωστή και ισόρροπη των περιφερειών της είναι απαραίτητη για να προχωρήσει και η ανταγωνιστικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να πετύχουμε τους στόχους της 2020. Είναι πολύ σημαντική λοιπόν γιατί δημιουργεί θέσεις εργασίας, βελτιώνει τα δίκτυα μεταφορών. Νομίζω λοιπόν ότι λόγω όλων αυτών δεν είναι σωστό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιεί τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για να απειλήσει τα κράτη-μέλη τα οποία προσπαθούν να τηρήσουν τους στόχους, να πετύχουν μάλλον τους οικονομικούς στόχους που έχουν αναλάβει την υποχρέωση να πετύχουν. Στην ουσία φύγετε με τα μέτρα σας ε, τις χώρες που έχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Ευχαριστώ κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να επισημάνω το εξής. Όταν μιλάμε για σύνοχη και κοινωνικά ζητήματα, εγώ δεν μπορώ να εξηγήσω στους ψηφοφόρους μου πως ε, εμείς αποφασίζουμε αυτά τα πράγματα όταν αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι που μετά την ένταξη έχει γίνει χειρότερη η ζωή τους. Μιλάω για τη Λετωνία. 34% του πληθυσμού αυτή τη στιγμή είναι φτωχοί. του πληθυσμού των συνταξιούχων έχει αυτές τις ελάχιστες ε, συντάξεις δεν είναι δυνατόν. Πρέπει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο η κοινωνική πτυχή. Εδώ πέρα μιλάμε για περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς και ανταγωνιστικότητα, δηλαδή το αντίθετο. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριος Γιά, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θέλω να κάνω τέσσερις παρατηρήσεις για τις εκθέσεις, κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι λογική για τους ανθρώπους μόνο εάν βελτιώνει και μειώνει τις κοινωνικές, οικονομικές και περιφερειακές ανισότητες. Δεύτερον, η πολιτική συνοχή είναι αποφασιστική σημασία μέσω για να πραγματοποιηθούν αυτοί οι στόχοι. Τρίτον, θα πρέπει να υπάρξει μια είτε μια εναλλακτική διατύπωση πρόταση, είτε καλύτερα όσοι την κακολογούν να μην λένε τίποτα. Τέταρτον, προέρχομαι από την Ανατολική Γερμανία. Έχουμε σημειώσει μεγάλε πρόοδου, αλλά ακόμα δεν τα έχουμε καταφέρει. Γι' αυτό χρειαζόμαστε και περαιτέρω υποστήριξη μετά το 2013 για να μπορέσουμε να παραμείνουμε στη σωστή πορεία. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ, κύριο Σεσόν Κέλλη, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εν συντομία, Θέλω να πω ότι ο Τίπο Νίλ, ένας μεγάλος Ρολανδός ε, ο πολιτικός, είχε πει ότι η πολιτική είναι τοπική, σε τοπικό επίπεδο και ότι θα μπορούσαμε να πούμε και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την ανάπτυξη. Η ανάπτυξη είναι περιφερειακή. Και στο πλαίσιο της ε, πολιτικής συνοχής νομίζω ότι η επιτυχία της χώρας μου είναι το τέλειο παράδειγμα σε ό,τι αφορά ε, το ΑΕΠ έχει αυξηθεί κατά 1,5% από το 1973 μέχρι σήμερα παρά τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Πρέπει να πω επίσης ότι για να προχωρήσουμε ε, μια σημαντική πτυχή θα είναι να απλωστεύσουμε τις διαδικασίες και να δώσουμε έμφαση στα αποτελέσματα, στην προσθέμενη αξία. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να περιστήλουμε τη γραφειοκρατία και τις ρυθμίσεις Εάν δεν υπάρχει προστιθέμενη αξία, δεν έχει καμία πρόοδο το να κάνουμε τίποτα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ολοκληρώσουμε το γύρο των ομιλητών αυτό με τον κύριο Μικολάσικ. Gracias, señor efektívne uplatňovanie politiky súdržnosti ktoré je v súčasnosti. η πολιτική συνοχή αγαπητέ κύριε πρόεδρε πρέπει να είναι μια πολιτική καταρχά απο, ε, μη συγκεντρωτική αποκεντρωμένη σε βάθο. τότε μόνο θα είναι χρήσιμη ε, προ τι ε, τοπικέ και περιφερειακέ, αρχέ, οι οποίε γνωρίζουν τι πραγματικέ ανάγκε του πληθυσμού του πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια σωστή εταιρική σχέση πριν από οτιδήποτε άλλο με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Αυτό σημαίνει πριν από οτιδήποτε άλλο ότι πρέπει να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, πρέπει να υπάρξει σωστό συντονισμός στις διαδικασίες ελέγχου και πρέπει να υπάρξουν διαδικασίες πολύ πιο ε, διαφανείς από ό,τι μέχρι σήμερα. Ευχαριστώ συνάδελφο. Ολοκληρώθηκε λοιπόν και η διαδικασία προσέλκυση τη προσοχή του Προέδρου. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Επίτροπο, τον κύριο Χάν, για να απαντήσει εκ μέρους τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, στις διάφορες παρεμβάσεις. Ευχαριστώ. Έχετε το λόγο κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ για τη συζήτηση αυτή και όπως είπα, να το με τις να πω κάποια πράγματα για τον έλεγχο. Αυτό οπωσδήποτε, και το λέω πάντα, είναι ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει, να γίνουν τα πράγματα απλούστερα, ειδικά δεδομένου του ότι ε, πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο να δώσουμε τη δυνατότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν τα ευρωπαϊκά ταμεία. Και να έχουμε τα μία τρέχοντα ας πούμε τα οποία συνεχώς θα είναι σε λειτουργία και να μειωθεί οπωσδήποτε η γραφειοκρατία. Βεβαίως ένα μεγάλο κομμάτι της γραφειοκρατίας προστίθεται σε εθνικό επίπεδο. Δηλαδή ό,τι βλέπετε στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού έργους γραφειοκρατία δεν προέρχεται από τις Βρυξέλλες είναι το σύνολο, εάν θέλετε, εθνικών και ευρωπαϊκών πρωτεγραφών. Και πράγματι, όπως είπε η κυρία Μανέσκου, πρέπει να αναπτύξουμε κάποιες πρωτεγραφές, αλλά δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε τελείως τις εθνικές νομοθεσίες και ιδιαιτερότητες, αλλά επί της αρχής συμφωνώ. Επίσης το θέμα της αιρεσιμότητας. για το οποίο δεν μπορούμε να αφιερώσουμε τόσο χρόνο όσο θα θέλαμε, αλλά για κάθε χώρα και για κάθε περιφέρεια θα πρέπει να βρούμε τους λόγους και συχνά τους ξέρουμε για τους οποίους υπάρχουν καθυστερήσεις στην εφαρμογή των έργων. Συχνά αυτό δεν έχει καμία σχέση με τα λεφτά, αλλά με άλλα, άλλες ελλείψεις. Αυτές θα πρέπει να αντιμετωπιστούν εκ των προτέρων προς το συμφέρον όλων των ε, ενδιαφερομένων. Εκεί πέρα αυτό είναι το σκεπτικό, αν θέλετε, των όρων αυτών της αιρεσιμότητας. Επίσης, σας ευχαριστώ για αυτό το οποίο είπατε για την σύμβαση αυτή της ανάπτυξης και της εταιρική ε, σχέσης ε, και ο κ. Όλμπριχτ είπε πως θα πρέπει να δούμε την ε, συνεισφορά τοπικού και περιφερειακού επίπεδου. Εδώ πέρα πρέπει να επανεξετάσουμε τα πράγματα, να δούμε πώς θα μπορέσουμε να δούμε τι θα κάνουμε με την εφαρμογή και κάτι το οποίο πρέπει να αποδεχθούν, κάτι το οποίο πρέπει να αποδεχθούν και τα κρατημέλη και γι' αυτό εδώ πέρα θέλω τη στήριξη του Κοινοβουλίου γιατί όπως ξέρετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι στο πλευρό μας υπάρχει βεβαίως και η Επιτροπή των Περιφερειών αλλά υπάρχει και ο βασικότερος παίκτη που είναι εδώ πέρα τα κράτη-μέλη τα οποία πρέπει να πείσουμε αλλά πρέπει να τα πείσουμε πως υπάρχει και μια προστιθέμενη αξία όταν ασχολούνται περισσότεροι άνθρωποι με τον προγραμματισμό των ε, προγραμμάτων αυτών και θα μπορέσουν να δουν τυχόν ελλείψεις. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Ε, ε, άκουσα κάποιες δηλώσεις νομίζω των πρασίνων που μίλησαν για την ανάπτυξη. Αν είναι σωστό το να έχουμε όλο περισσότερα. Εγώ είμαι υπέρ και της ποσοτικής και της ποιοτικής ανάπτυξης. Και τα δύο χρειαζόμαστε. Και αν σκεφτούμε την έρευνα, νομίζω κατ' ουσίαν ανήκει στην κατηγορία της ποιοτικής ανάπτυξης. Π.χ. ένας από τους μεγαλύτερους στόχους μας είναι η αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά ταυτόχρονα να έχουμε και μεγαλύτερη αποδοτικότητα τη ενέργειας. Οπότε το θέμα της έρευνας είναι πώς θα μπορέσουμε να αποθηκεύσουμε, μεταφέρουμε και διαθέσουμε τον ηλεκτρισμό όταν τον χρειαζόμαστε. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για να είμαστε ακόμη πιο αποτελεσματικοί στην παραγωγή ενέργειας. Γενικά, και νομίζω και αυτό ήταν σαφές, θα επιτύχουμε τους στόχους μόνο εάν έχουμε μια περιφερειακή πολιτική η οποία θα φτάσει σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης γιατί και αυτό κατέστη σαφές ότι δηλαδή εάν θέλουμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα του 2020. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο εάν μεταφερθεί αυτή η πολιτική σε όλες τις περιφέρειες, εφαρμοστεί εκεί πάντα σεβόμενη τις τοπικές ιδιαιτερότητες. Ευχαριστώ λοιπόν τους δύο για την εργασία τους. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ και θα δώσουμε τώρα το λόγο στους δύο Πρώτα απ' όλα στον κύριο Λούχαν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Α, ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους ε, που συνεισέφεραν στη σύνταξη αυτής της έκθεσης για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Ευχαριστώ επίσης τους συναδέλφους εκείνους που συνεισέφεραν με τροπολογίες και μπορέσαμε έτσι τελικά να βρούμε ε, κάποια συνένεση. Θα ήθελα παρόλα αυτά να συμφωνήσω με αυτό το οποίο είπε και ο κύριος Επίτροπος, δηλαδή πως πολιτική συνοχή είναι πολιτική επένδυση στις περιφέρειες και πρέπει να είναι πολιτική επένδυση ε, στις περιφέρειες και τους ε, ανθρώπους ε, και να έχει στόχο την αύξηση των καλυτέρευση των συνθήκων ζωής σε όλες τις περιφέρειες. Σας ευχαριστώ λοιπόν που είστε στο πλευρό μας. Εμείς Συμφωνούμε επίσης πως ε, είναι σημαντική η επένδυση στις υποδομές για να καλυφθεί αυτή η διαφορά που υπάρχει αυτή τη στιγμή μεταξύ περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά τώρα τον κύριο Μπεσέ, εάν είχε διαβάσει την έκθεση θα ήξερε πως ε, η έκθεση μιλάει και για ανάπτυξη ε, με σεβασμό στο περιβάλλον. Τα λέμε αυτά. Και μιλάμε για πράσινη οικονομία στην έκθεση. Ελπίζω η έκθεση να ικανοποιήσει την πλειοψηφία και ελπίζω έτσι να, έχει, να είναι σε καλό δρόμο το μέλλον της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής. Σας ευχαριστώ και θα ολοκληρώσουμε με την παρέμβαση της δεύτερης της κυρίας εισηγήτριας Μανέσκου που έχει πει δύο λεπτά για την παρέμβασή της. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την συνεισφορά τους στην τελική μορφή της έκθεσης. Ευχαριστώ για όλες τις βελτιώσεις, ευχαριστώ για τις συνεισφορές στη συζήτηση απόψε με την ε, ψηφοφορία στην Επιτροπή Περιφερειακών ε, Θεμάτων ε, φάνηκε πως υπάρχει υποστήριξη για αυτή την έκθεση για τα μέτρα τα οποία προτείνει και νομίζω χαίρομαι και για την απόψινή συζήτηση. Το έγγραφο εργασία το διαβουλευτήκαμε με την Επιτροπή των Περιφερειών, με την Κομισιόν και με τους εκπροσώπους των Περιφερειών. Σας ευχαριστώ όλους λοιπόν και όπως είπα και στην αρχή της συζήτησης, είμαι πεπισμένη πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι αποφασισμένη να εφαρμόσει τις λύσεις τις οποίες εμείς διατυπώσαμε στην Επιτροπή Περιφερειακών Υποθέσεων για να γίνουν πραγματικότητα οι προτάσεις μας. Τους επόμενους μήνες η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποφασίσει την μελλοντική πολιτική συνοχή στο πλαίσιο της ε, στρατηγικής 2020 για να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους. Πράγματι, επιθυμούμε να έχουμε ορθή διακυβέρνηση σε πολλά επίπεδα τη λεγόμενη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση έτσι ώστε να έχουμε και κοινωνική πρόοδο και πιο αηφόρο ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Ολοκληρώθηκε σημαντική αυτή η συζήτηση. Η ψηφοφορία του αντίστοιχου ψηφίσματος θα λάβει χώρα αύριο στις 12 το μεσημέρι. Και τώρα περνάμε στο επόμενο σημείο της μερισιάς διάταξης που είναι η έκθεση του συναδέλφου μας Φιλίπ Ζουβά με θέμα τον αντίκτυπο της διαφήμισης στη συμπεριφορά των καταναλωτών. Όπως γνωρίζετε, η διαδικασία στη συζήτηση αυτή είναι ότι μετά την παρέμβαση